fratelli. Bene, benvenuti a tutti. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Σας καλωσορίζω όλους, επαναλαμβάνει ο κ. Δεκάστρο. Είναι χαρά μου να κηρύξω την έναρξη αυτής της συνεδρίασης για την εκ νέου δραστηριοποίηση της ένατης κοινοβουλευτικής περίοδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Έχουμε μπροστά μας αποφασιστικές θα έλεγα προκλήσεις ε, και μόνο ενωμένοι στο Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να προασπιστούμε την γεωργία και τα 10 εκατομμύρια των γεωργών όπως και τα 500 εκατομμύρια των καταναλωτών στην Ευρώπη. Να σας θυμίσω ότι ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας, υπάρχουν 22 γλώσσες στην διερμηνία εκτός από τα ε, κέλτικα και τα μαλτέζικα. Αποκλειστικό στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή του, η εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Θα πρέπει να ψηφίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Αν έχετε ξεχάσει την κάρτα σας, υπάρχουν προς αντικατάσταση κάρτες στους κλητήρες. Πρέπει να ελέγξετε αν έχετε όλη την κάρτα σας θα περάσουμε πρώτα στην εκλογή του νέου Προέδρου και μετά θα περάσουμε στην εκλογή των τεσσάρων αντιπροέδρων, σύμφωνα με τον κανονισμό. Η απαραίτητη απαρτία για την εκλογή του Προέδρου μας είναι 12 μέλη τα οποία πρέπει να παρίστανται. Ο μέγιστος αριθμός των ψήφων είναι 48. Οι αναπληρωτές που είναι παρόντες σήμερα εφόσον απουσιάζουν τα πλήρη μέλη πρέπει να μας το πούν. Α, έχουμε ήδη τα ονόματα λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Έχουμε κάποιους αναπληρωτές. Σαββαμά, Μπρέντφορτ, Εγώ αντικαθιστώ τον Μπράτφορντ. Ο κύριος Λεμπρετό αντικαθίσταται από την κυρία Μέλη. Και οι Ντότς αντικαθίστανται επίσης από τον κύριο Σίντσι. Καλώς. Ο Ξεχάσατε να αναφέρετε το δικό μου όνομα. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Σαβαρμά. Πέτερ Γιάρ, για τα πρακτικά. Okay. Εντάξει, λείπει ο Σαβαρμά που αναφέρατε το όνομά του, εγώ τον αντικαθιστώ. Ναι, ξέχασα να πω το όνομά σα. Είπα ότι θα αντικατασταθεί ο κύριο Πέτρη Σαβάρμα, αλλά δεν είπα ότι αντικαθίσταται από εσά. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργεί σωστά το ηλεκτρονικό σύστημα και αυτό θα μας δώσει και τη διαβεβαίωση ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί σας. Αν είστε όλοι έτοιμοι, δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Είπαμε είναι μια απλή δοκιμή. Έχουμε ένα μέλος των σοσιαλιστών επιπλέον. Ο Μάρκ Ταραμπελά. Μην κάνετε κόλπα. Πάλι υπάρχει μία ψήφος επιπλέον σοσιαλιστές. θα πρέπει να είμαστε 48 αλλά είμαστε 49. Βέβαια η μηχανή δεν μας λέει ποιος είναι ο επιπλέον, ποιος είναι ο 49ος. Μόνο τα πλήρη μέλη και οι αναπληρωτές τους οποίους προαναφέραμε. Κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Τώρα είμαστε 48. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση. Ο κύριος Ατσόλος δεν είναι εδώ και θέλουμε να ψηφίσουμε τον Σαλς Κιόρενς. Εφτά δηλαδή ε, θα είμαστε εμείς. Okay, We will take notes about that. Θα το σημειώσουμε, εντάξει. Oh. Ai relatori dei gruppi politici θα ζητήσω τώρα από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να ανακοινώσουν τους υποψηφίους τους για τις θέσεις πρώτα του Προέδρου. Να σας θυμίσω ότι κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι πλήρες μέλος. Θα πρέπει να έχει συμπληρώσει πλήρως την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την δήλωση σεβασμού του κώδικα συμπεριφοράς. Λοιπόν, οι πολιτικές ομάδες. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η ομάδα ID Σας παρουσιάζουμε την υποψήφια. Η κυρία Μαξέτ Πιμπαρκάς. Δέχεστε την πρόταση για την υποψηφιότητά σας. Ναι, δέχομαι την πρόταση, λέει η κυρία Πιμπάρκας. Ευχαριστώ. Οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σαν συντονιστής του συγκεκριμένου κόμματος στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρο θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τον κύριο Νόμπεν Λίντς υποψήφιο πρόεδρο. accetta Κύριε Λίντς, δέχεστε την υποψηφιότητα. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, επιβεβαιώνω ότι η κυρία Μαξέντ Πιμπαρκάς και ο κύριος Λίντς είναι πλήρη μέλη, έχουν συμπληρώσει πλήρως τις δηλώσεις δημοσίου οικονομικού μάλλον συμφέροντος, όπως επίσης και έχουν υπογράψει και τον κώδικα συμπεριφοράς και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ εδώ να με προσέξετε. Για να ψηφίσετε για τον κύριο Λίντς θα πρέπει να πατήσετε το κόκκινο κουμπί. Και για να ψηφίσετε για την κυρία Πιμπαρκάς θα πρέπει να πατήσετε το πράσινο κουμπί. Εντάξει. Λοιπόν, μία ψηφοφορία θα γίνει για τον υποψήφιο του ΕΛΚ θα πατήσετε το κόκκινο και για να ψηφίσετε την κυρία Πιμπάρκας του ID θα πρέπει να, ψηφίσετε, να πατήσετε το πράσινο. Νομίζω ότι είναι σαφές. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ο κύριος Λίντς πήρε 36 ψήφους και η κυρία Πιμπάρκας 11 ψήφους. Συνεπώς ανακηρύσω τον κύριο Λίντς ως πρόεδρο της Επιτροπής μας. Πήρε την απόλυτη πλειοψηφία και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να αναλάβετε πλέον την Προεδρία μας. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη σας. Πιστεύω ότι μας περιμένει πολλή δουλειά με τη γεωργική μεταρρύθμιση και όλα τα άλλα θέματα που απασχολούν τους αγρότες και τις αγρότησες Ευρώπη, αλλά και περιμένουν από εμά, όπως και οι καταναλωτές και οι καταναλώτριοι. Και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αρχίσουμε δουλειά. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, συγκρότηση της Επιτροπής μας σε σώμα και να προχωρήσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. Άρα, θα μιλήσω αγγλικά για να μην γίνει κανένα λάθο. Και θα σα αναγνώσω όλα αυτά που μας περιμένουν. Από ε, αρχαιρεσίε. Προχωρούμε λοιπόν στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής Άγκρη, Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου και μετά ξεχωριστά και διαδοχικά θα προχωρήσουμε στην εκλογή του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου αντιπροέδρου. Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό η απαρτία που απαιτείται για την εκλογή των διαφορών αντιπροέδρων είναι 12 μέλη. Και ο μέγιστο αριθμό μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν είναι 48, είτε πρόκειται για τακτικά μέλη είτε για αναπληρωματικά. οι παρόντες αναπληρωτές είναι γνωστοί, δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσουμε το κατάλογο. Αν θέλουν να αλλάξουν τους αναπληρωτές, ε, οι διάφορες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το δηλώσουν πριν την ψηφοφορία, αλλά δεν νομίζω να ζητεί κανείς το λόγο. Ε, κύριε Μελά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για λόγους σεβασμού της δημοκρατίας και της πολυφωνίας στο θεσμικό μας όργανο, η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία θα ήθελε να καταθέσει την υποψηφιότητα της κυρίας Μαξέτ Πιμπαρκάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο de la première... Για πρώτη αντιπρόεδρο. Δεν ξέρω αν το είπα λάθος. Ωραία. Καλώς. Τώρα όμως δεν είχαμε φτάσει ακόμα στις υποψηφιότητες, αλλά δεν πειράζει. Σημειώνουμε την υποψηφιότητα αυτή. Προχωρώ. <laughs> Ήθελα επίσης να θυμίσω ε, ότι θα πρέπει να αντανακλάται στη σύνθεση του Προεδρείου η γεωγραφική ισορροπία και η ισορροπία του φύλου. Παρακαλώ τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να δηλώσουν τις υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής μας και να έχει υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, καθώς επίσης και τη δήλωση ε, σεβασμού του κώδικα ε, διοντολογίας και συμπεριφοράς. Έχουμε υποψηφιότητες. Ο Μάρτιν Χόισλεγκ. Προτείνω τον Φρανσίσκο Κεγέρο για πρώτο αντιπρόεδρο. Ο Φρανσίσκο Γκερέρο προτείνεται. Η ομάδα ID πρότεινε την κυρία... And, uh, uh, Την κυρία Πιμπαρκάς. Δέχεστε και οι δύο υποψήφοι την υποψηφιότητά σας. Την αποδέχεστε. Yeah. Oui, bien sûr, j'accepte la candidature. Βεβαίως και οι δύο. So, dann stellt sich die Frage, ob... Λοιπόν- Οπότε, να κάνουμε μυστική ψηφοφορία. Αυτό γίνεται όταν έχουμε Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα γίνει ούτω ή άλλω μυστική ψηφοφορία για, πρώτη, για, τον πρώτο αντιπρόεδρο. <clears throat> Λοιπόν, μυστική ψηφοφορία. Όποιο θέλει να ψηφίσει τον κύριο Γκερέρο θα πατήσει το πράσινο κουμπάκι. Όποιο θέλει να ψηφίσει την κυρία Πίμπαρκας θα πατήσει το κόκκινο κουμπάκι. Οπότε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. So, dann kann ich die. Where can I see? Yeah. Yeah. Dann kann ich die Abstimmung schließen. Πέρα τη ψηφοφορία. Για τον κύριο Γκερέρο έχουμε 38 ψήφους και για την κυρία Τιμπαρκάς 6. Κύριε Γκερέρο, παρακαλώ να έρθετε εδώ επάνω στο Προεδρείο. Συγχαρητήρια. Πάμε λοιπόν τώρα στον δεύτερο ή στην δεύτερη αντιπρόεδρο. Υπάρχουν προτάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καταθέτω Ευχαριστούμε την υποψηφιότητα του κυρίου Ντανιέλ Μπούντα για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου της Επιτροπής Γεωργίας. Άλλε weitere Άλλες προτάσεις υπάρχουν? Παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω, πάντα ε, ε, υπέρ του σεβασμού της πολυφωνίας και της δημοκρατίας η ομάδα μας ε, καταθέτει την υποψηφιότητα της κυρίας Μαξέτ Πυρμπακάς για τη θέση του δευτέρου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άλλες προτάσεις, άλλες υποψηφιότητες. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, πάμε πάλι στην ψηφοφορία. Όποιος θέλει να ψηφίσει τον κύριο Μπούντα θα πατήσει το πράσινο κουμπί. Όποιος θέλει να ψηφίσει την κυρία Πύρμπακας θα, θα πατήσει το κόκκινο κουμπί και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Dann können wir die Abstimmung abschließen. Πέρας της ψηφοφορίας. Για τον συνάδελφο Μπούντα έχουν ψηφίσει 37 άτομα, για την κυρία Πύρμπακας 7. Κύριε Μπούντα, παρακαλώ να έρθετε εδώ στο Προεδρείο. <clears throat> Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, για τις επόμενες δύο ψηφοφορίες μάλλον θα υπάρξουν δυσκολίες. Mm. Γι' αυτό έχουν ζητήσει διάφορες ομάδες να πάρουν το λόγο. Θα το επιτρέψω. Και ελπίζω βεβαίω να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα χρονοδιαγράμματα γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε και από την αίθουσα σύντομα. Ποιο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Νομίζω ότι να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλέρ και συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι τώρα πρόκειται για τον τρίτο αντιπρόεδρο, όπου υπάρχουν πολλοί υποψήφοι και θα παρακαλούσα όμως ε, να προχωρήσουμε στην εκλογή του τετάρτου αντιπρόεδρου, που δεν είναι επίμαχη για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια ε, έτσι, για τους συναδέλφους να ψηφίσουμε πρώτα για τον τέταρτο αντιπρόεδρο και την άλλη φορά για τον τρίτο. Ο κύριος Χόισλινγκ, συμφωνώ με την κυρία Μίλλερ να ψηφίσουμε για τον τέταρτο αντιπρόεδρο, προλαβαίνουμε και να αναβάλουμε την ε, εκλογή του τρίτου αντιπρόεδρου. Okay. Oh. It's me. Thank ECR e Εξ ονόματος της ομάδας ECR θα ήθελα να προτείνω για τη θέση ε, του τετάρτου διπρόεδρου την κυρία Μαζολία Αγγιλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αμελέ, νομίζω ότι οι καλοί τρόποι επιβάλλουν για να στείλουμε και ένα καλό μήνυμα ε, να μην αναβάλουμε την ε, εκλογή του τρίτου ή της τρίτης αντιπροέδρου. Ζητώ να γίνει πάρα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ich glaube, dass wir jetzt über das Verfahren Λοιπόν, Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε λίγο την όλη διαδικασία. Υπάρχουν δύο αιτήματα για να μετατεθεί η ψηφοφορία. Καταρχάς να μεταθέσουμε τελείως τον τρίτο αντιπρόεδρο και τον τέταρτο, τις δύο αυτές εκλογές και υπάρχει το αίτημα δύο πολιτικών ομάδων να ψηφίσουμε τον τέταρτο ή την τέταρτη αντιπρόεδρο και να μεταθέσουμε μόνο την ψηφοφορία του τρίτου. οπότε να δούμε τώρα πού βρίσκεται η πλειοψηφία. Δύο ομάδες έχουν προτείνει να ψηφίσουμε τον τέταρτο αντιπρόεδρο και οι σοσιαλιστές προτείνουν και τις δύο αυτές τι πληροφορίε για τον τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο να τις μεταθέσουμε. Οπότε προτείνω ένα λεπτό. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι να ψηφίσουμε τον τέταρτο πρόεδρο τώρα. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Ναι, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Αλλά αν δεν ψηφίσουμε τον τρίτο αντιπρόεδρο, μάλλον πρέπει να κλείσουμε εδώ τη συνεδρίαση και να περιμένουμε μέχρι την ε, επόμενη συνεδρίαση. Ούτως ή άλλως στις επόμενες δύο εβδομάδες δεν πρόκειται να γίνει κάτι και μετά να συνεχίσουμε με τη σωστή σειρά της ψηφοφορίας. Να ψηφίσουμε δηλαδή πρώτα τον τρίτο και μετά, έτσι όπως λένε και οι κανόνες. Τον τέταρτο. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία να ακολουθήσουμε. Αν τώρα κάνουμε μετάθεση, θα πρέπει να μεταθέσουμε και τις δύο ψηφοφορίες. Και μετά σε δύο εβδομάδες να ψηφίσουμε και τους δύο εναπομείναντες αντιπρόεδρους. Εντάξει. Οπότε, η πρόταση τώρα είναι και οι δύο εναπομείναντες ψηφοφορίες να μετατεθούν. Ποιος συμφωνεί, παρακαλώ, δια της άρσεως της χειρός. Okay. Ωραία. Καλύτερα να το δούμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ποιο είναι υπέρ τη παράταση των αντιπροέδρων 3 και 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Όποιο είναι υπέρ ψηφίζει πράσινο. Όποιο είναι αντίθετο, ψηφίζει κόκκινο. Okay, dann schließe ich die Abstimmung. Ωραία. 29 λοιπόν ψήφοι υπέρ της, της μετάθεσης και 16 κατά. Επομένως θα ψηφίσουμε στις 23 Ιουλίου τον τρίτο και τον τέταρτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Το μόνο που έχω να πω για το τέλος της συνεδρίασης είναι να σας πω πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση. Είναι στις 23 Ιουλίου ...23 Ιουλίου το πρωί και το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους. Και μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίαση.